του κυρίου Όλι Ρεν που απεχώρησε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών λήγει την Τρίτη στις 6 το απόγευμα. Οι υποψηφιότητες πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο του Γενικού Γραμματέως της ε, Προεδρίας, στο γραφείο ΡΟ 00101, στην Espace Paysager de la Présidence, στο ε, κτίριο Louis Weiss, Εκεί λοιπόν μπορούν να κατεθούν οι υποψηφιότητες και η δήλωση αποδοχής πρέπει να προσθεθεί, να συμπληρώνεται και αυτή.